ψηφοφορίε τώρα. Ξεκινούμε με την έκθεση Γκρόμπαρτσικ σε σχέση με τα αποθέματα Σολομού στην Βαλτική. Υπάρχει μονάχα μία ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Πέρας ψηφοφορίας. γίνεται δεκτή η έκθεση. Ακολουθεί η έκθεση Lightfried για τις αρμοδιότητες που αφορούν ορισμένα μέτρα εμπορικής πολιτικής και πάλι είναι μόνο μία ψηφοφορία ονομαστικού χαρακτήρα άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Γίνεται δεκτή η έκθεση. Ερχόμαστε στην έκθεση του κυρίου Γκάλαχερ για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων. Ο κ. Γκάλαγκερ για διαδικαστικό θέμα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα εκτιμούσα ιδιαίτερα αν δεχόσασταν, ακόμα και αν είναι κάπως καθυστερημένο, να δεχτείτε την αίτησή μου για μια ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 32 και την τροποποιημένη πρόταση. Ο αποχρόν λόγος θα γίνει σαφής όσο προχωρούμε. Μάλιστα. Μπλοκ 1, τροπολογία 32 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία 32 και ερχόμαστε και το δεύτερο μπλοκ εκπίπτει. Ψηφίζουμε το κείμενο πώς έχει τροποποιηθεί. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Πέρασε ψηφοφορία. Γίνεται δεκτό το τροποποιημένο κείμενο. Ερχόμαστε στην τροπολογία 33 ο κύριος Γκάλαχερ. Παρακαλώ κύριε Γκάλαχερ. Α, τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κύριε, κύριε Γκάλαχερ, παρακαλώ. Η Επιτροπή Αλληλείας θεωρεί πως ε, ως ε, κοινοβούλιο δεν έχουμε άλλη εναλλακτική παρά να καταδικάσουμε την ε, στάση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλληλείας. Διαδοχικές προεδρίες αγνόησαν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη τα τελευταία τρία χρόνια για ζητήματα που αφορούν τα πολυετή σχέδια. Τα πολιετή σχέδια είναι ο πυλώνας της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και είναι πάρα πολύ σημαντικά για την προστασία των αλλιευτικών πόρων και για την διασφάλιση της επιβίωσης των αλλιευτικών κοινοτήτων. Εμείς λοιπόν ως το ερετό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε κοινή ευθύνη με το Συμβούλιο Υπουργών ως συνομοθέτες. Το Συμβούλιο Υπουργών πρέπει να αντιληφθεί τις ευθύνες αυτές και να σεβαστεί τη συνθήκη της Λισαβόνας και τους πολίτες της Ένωσης. Εξ ονόματος λοιπόν της Επιτροπής Αλίας ζητώ να αναβληθεί η τελική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο 1774 του κανονισμού και ελπίζουμε αυτή να είναι η πρώτη φορά και να ακολουθήσουν και άλλες για να αναγκάσουμε το Συμβούλιο να ε, έρθει μαζί μας σε ουσιαστικές συνομιλίες για αυτή τη διαφωνία που συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια. Έχει ζητηθεί αναβολή. Ποιος συμφωνεί με αυτήν. Κατά. Αποχές. Δεκτό το αίτημα. Περνάμε στην έκθεση Πατράου Νέβες Κυρία Αντζελίλη. Πρόεδρε, δέκα δευτερόλεπτα για αυτήν την έκθεση έχει διανεμηθεί αυτό εδώ το παιχνιδάκι. Είναι ένα κουκλάκι που ε, απεικονίζει ένα καρχαρία και το κοινοβούλιο όμως ξέρουμε ότι έκανε πάρα πολλά για την ασφάλεια και αυτό το καρχαριάκι εδώ δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές. Γι' αυτό λοιπόν κακό, καλό είναι να μην κυκλοφορούν παρόμοια προϊόντα για την επικίνδυνα για την υγεία. Κυρία Αντζελίλη, και αυτή η τοποθέτηση ήταν σημαντική, αλλά δεν ήταν επί της διαδικασίας. Άλλη φορά θα διακόπτω όποιον δεν ασχολείται με ζητήματα ε, διαδικαστικά. Παρακαλώ. Πρόεδρε, να πω στους συναδέλφους ότι Επιστροπολογία 14 της ε, λόγω έκθεσης στον κατάλογο των ψηφοφοριών υπάρχει ένα πλήν, ενώ θα έπρεπε να είναι θετικό. Ένα λάθος λοιπόν έχει επισέλθει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση Πατράων. Εύε αφαίρεση, πτερυγείο, καρχαρία, επί του σκάφου. 11 τροπολογίες πρώτα της Επιτροπής υπέρ κατά Το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορία έχει αποσυρθεί. Ποιος είναι υπέρ των 11 τροπολογιών της Επιτροπής. Κατά. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτές. Τροπολογία 14 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή η 9 έχει καταπέσει. Τροπολογία 18 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Οπότε οι τροπολογίες 8, 15, 16, 17 έχουν καταπέσει. Ψηφίζουμε την πρόταση όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά Θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Με ναι, σαφή πλειοψηφία. Κοιτάξτε, πριν είδα αλλιώ τα χέρια. Περνάμε στο ε, νομοθετικό ψήφισμα με νομοστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. δεκτό. Περνάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία για τη Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα διεθνούς απαγωγής παιδιών. Έχουμε ψήφισμα της Επιτροπής Νομικών παράγραφος 1 ε, δεκάρχη της ψηφοφορία, μονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. δεκτό. Εκτιμώντας G ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας H υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας I ποιο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Εκτιμώντας J υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό όλο το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε τώρα σε τρία ε, νομοθετικά ψηφίσματα που αφορούν την παγκόσμια διάσκεψη για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες. Έχουμε πρώτα απ' όλα πρόταση τεσσάρων ομάδων. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία αυτή. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το ψήσιμο σύνολό του υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για, για ζητήματα περιβάλλοντος, ε, έτοιμα 8 με συγχωρείτε, πολιτικών ομάδων. Πάρκο 7 σε τρία μέρη. μέρο πρώτο υπέρ, κατά, αποχέ δεκτό. Δεύτερο μέρο υπέρ, κατά, αποχέ δεκτό. Τρίτο μέρο υπέρ, κατά, απόχέ, δεκτό. Παράγραφος 8 σε δύο μέρη. Μέρο πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο μέρο υπέρ, κατά, αποχές δεκτό παραγραφός 9 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό παραγραφός 11 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 12 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 22. μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 21 ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτό. Παράγραφος 22, το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 28, σε δύο μέρη, με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται τη ψηφοφορία για το πρώτο μέρος. Ψησαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Επίσης ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Ε, επίσης συγκρίνεται. Παράγραφος 29 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παράγραφος 36 το αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Παραγραφός 37 το αρχικό κείμενο. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα το επαληθεύσουμε όμως ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 3. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 43 το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Παραγραφός 43. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παράγραφος 44, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 51, σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 63. Αρχικό κείμενο σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος τρίτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 66 το αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μετά την παράγραφο 73 περνάμε στην τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 77 τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 77 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές δεκτό μετά την παράγραφο 79 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή Παράγραφος 82 αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Παράγραφος 83 μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Το ψήφισμα στο σύνολό του άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Δεκτό. Ερχόμαστε στην έκθεση ΚΟΠΑ, διεύρυνση πολιτικέ κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγραφος 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Δεκτό δεύτερο τμήμα. Παράγραφο 26. Αρχικό τμήμα. Πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 27 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Παράγραφος 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές κάνουμε έλεγχο ηλεκτρονικό άρχεται η ψηφοφορία ψήφισατε όλοι πέρας γίνεται δεκτό και αυτό το τμήμα παράφος 38 του αρχικού κειμένου με χωριστή ψηφοφορία ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο ως με ονομαστική κλίση, το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Γίνεται δεκτό το ψήφισμα. Ακολουθεί η ψήφιση 7 ψηφισμάτων για την κατάσταση στη Γάζα. Καταρχήν αυτό το ψήφισμα των 5 πολιτικών ομάδων. Η κυρία Ντεκάιζερ, θέλετε να λάβετε το λόγο για να κάνετε μια προφορική τροποποίηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λόγω της κατάπαυσης πυρός που έλαβε χώρα χθες στην Γάζα, θέλουμε να τροποποιήσουμε, με τη συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων, την διατύπωση και υπάρχουν τέσσερις προφορικές τροπολογίες που θα σας αναφέρω καθώς προχωρούμε. Μπορώ να σας αναφέρω την πρώτη ε, προφορική τροποποίηση στην αρχή της παραγράφου 1 εκφράσει τη βαθιά ανησυχία λοιπά. Υπάρχει η προστίκη, χαιρετίζει την ε, κατάπαυση του πυρός και ε, καλεί για την πλήρη εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός. Και ε, εκφράσει την ικανοποίησή τη για την, την ικανοποίησή του κοινοβούλου για τι προσπάθειε τη Αιγύπτου για την επίτευξη τη κατάπαυση του πυρό. Θέλετε να σα διαβάσω όλη την παράγραφο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεκάιζερ. Υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική αυτή τροποποίηση στην παράγραφο 1. Εάν όχι, ψηφίζουμε ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2, τροπολογία 1, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Ψήφι 5. παραγράφω 7. Κατά. Αποχές δεκτή. Αιτιολογική σκέψη μετά την παράγραφο 4, κυρία Ντεκάζερ έχει το λόγο. Θα σας διαβάσω και τις τρεις προφορικές τροποποιήσεις. Μια νέα αιτιολογική σκέψη, λαμβάνοντας υπόψη την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός της 21ης Νοεμβρίου 2012, η δεύτερη τροπολογία δεδομένου του ότι η πρόσφατη κλιμάκωση βίας έχει οδηγήσει σε απώλεια, σε απώλεια ζωής και όχι η συνεχιζόμενη σύραξη και η τρίτη, η τέταρτη τροπολογία στα αγγλικά ζητώ συγγνώμη για τους Βρετανούς συναδέλφους τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά δεδομένου ότι ο Καμέλα, υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου και η υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρη Κλίντον, ανακοίνωσαν σε μία συνέντευξη τύπου στο Κάιρο την κατάπαυση πυρός στις 21 Νοεμβρίου 2012 δεδομένου ότι βάσει αυτής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός το Ισραήλ θα πάυσει κάθε εχθροπραξία στη λόριδα της Γάζης από ξηρά θαλάσσης και αέρος και αυτό αφορά και την στόχευση συγκεκριμένων ατόμων αυτό είναι παράθεση από τη συνέντευξη τύπου και επίσης ότι όλες οι Παλαιστινιακές φατρίες θα σταματήσουν εχθροπαξίες κατευθυνόμενες από τη, από τη λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων με πυράβλους και επιθέσεις κατά μήκο της συνοριακής γραμμής και κλείνει εδώ πάλι η Αγγίλη. Πάλι πρόκειται για μια παράθεση από την συνέντευξη τύπου. Αυτή είναι η τροπολογία μου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβατε τις τρεις τροπολογίες της κυρίας Κάιζερ, ε, Kaiser, για την παραγραφό 4, για την αιτιολογική σκέψη Α. Επίσης, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για αυτές τις τρεις τροπολογίες, μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού για τις τρεις αυτές τροπολογίες. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Ούτως απεφασίστη. Το σύνολο του ψηφίσματος τώρα ψήφι κατά αποχές δεκτό το ψήφισμα. Περνάμε στην έκθεση Donjon για την εφαρμογή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας παράγραφος 1 τροπολογία 8 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 21 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Γίνεται δεκτή η παράγραφος 21. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν γίνεται δεκτή. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται επίσης. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές γίνεται δεκτή τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 παράγραφος 51 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Δεκτή. Παράγραφος 62. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και η παράγραφος 62 γίνεται δεκτή. Τροπολογία 19. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 101 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος ε, 108 Ποια Πέρας 102 συγγνώμη ναι. Δεκτή Τροπολογία 2 υπέρ Κατά Αποχές Απορρίπτεται Τροπολογία 3 υπέρ Κατά Αποχές Δεκτή Τροπολογία 4 υπέρ Κατά Αποχές Δεκτή το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας, δεκτή. Δεκτό το ψήφισμα. Ακολουθεί η έκθεση Πάσκου για την ρήτρα αμοιβαία άμυνα και αλληλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση. Παράγραφο 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 14. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό και το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 18 σε δύο τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Αιτιολογική σκέψη σίγμα τάφ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Το σύνολο όπως έχει τροποποιηθεί άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η έκθεση Κέλαμ ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνόχωρο. Μόνο μια συνολική ψηφοφορία ονομαστική, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έκθεση Τάραντ για το ρόλο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της κρίσης που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές. Τροπολογία 22 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 24. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έλεγχο στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου 20. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην παραγραφό 24 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κάνουμε έλεγχο για το δεύτερο τμήμα της 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. η ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Παράγραφος 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Δεκτό δεκτή η έκθεση. Ερχόμαστε στην έκθεση για κονσάρι. Διαπραγματεύσει για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας με το Καζακστάν. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μια προφορική ε, τροπολογία πιανού της κυρίας Γιακονσάρη, της εισηγήτριας. Παρακαλώ, κυρία Γιακονσάρη. Κύριε Πρόεδρε, Έχουμε μια προφορική τροποποίηση λόγω αρνητικών ειδήσεων από το Καζακστάν. Φαίνεται ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται στο Καζακστάν. Γι' αυτό η προφορική μου τροποποίηση που υποστηρίζεται από πολλές πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την βαθιά μας ανησυχία σε σχέση με την ε, δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε από τον εισαγγελέα Γενικό Εισαγγελέα του Καζακστάν κατά του κόμματος της αντιπολίτευσης και της ε, οργάνωσης Μέντια και ζητώντας την καταδίκη τους ως εξτρεμιστές και την απαγόρευση λειτουργίας αυτής της Ένωσης. Χρησιμοποιείται λοιπόν ο νόμο κατά τη τρομοκρατία και του εξτρεμισμού, αλλά θεωρούμε ότι αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για να καταστήλει τι διε... τις ενέργειες της αντιπολίτευσης και για να φημώσει την ελευθερία έκφραση. Ευχαριστώ πολύ. Λέω πρόεδρο, υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή προφορική τροποποίηση. Τροπο... Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 2 σε δύο τμήματα ψήφι υπέρ για το πρώτο τμήμα κατά δευ... αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η τροπολογία 3 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Δεκτή. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Έλεγχος για την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. πέρα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Α. Λατινικό. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. J ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Έλεγχος του πρώτου τμήματος της 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά. Ε, τροπολογία 1 υπέρ. 9 ε, ναι, με συγχωρείτε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται το ψήσιμο σύνολό του υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Περνάμε στην έκθεση Φεέρα Μικλή Κλίμακα Αλία και Παραδοσιακή Αλία και Μεταρρύθμιση τη Κοινή Αλληλευτική Πολιτική. Παράγραφο 3. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτή. Παράγραφος 31. Πρώτο εδάφιο σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παραγραφός 31 εδάφιο 3 σε 2 μέρη μέρο πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό. Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος της παραγράφου 31 τρίτο εδάφιο άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παραγραφός 31, τέταρτο εδάφιο, αρχικό κείμενο, μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παραγραφός 33 αρχικό κείμενο σε δύο μέρη υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 38 σε δύο μέρη αρχικό. Σε τρία μέρη. Αρχικό. Με πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό τρίτο μέρος με ονομαστική ψηφοφορία Άρχιτη ψηφοφορία Άρχιτη ψηφοφορία για το τρίτο μέρος ψήφισαν όλοι πέρας δεκτό Παράγραφος 40 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος πέρα κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας δεκτό εκτιμώντας ε σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά θα το επαληθεύσουμε άρχεται τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Angenommen. Δεκτό. Εκτιμώντας J. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Περνάμε τώρα στην έκθεση Λέβιν για εξωτερική διάσταση της κοινή αριευτικής πολιτικής. Τροπολογίες 1-8 έχουν αποσυρθεί. Περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Αρχικό κείμενο. Μέρος 1. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές θα το επαληθεύσουμε. Παραγραφός ένα δεύτερο μέρος ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παραγραφός 2 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 6 σε 2 μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παράγραφος 9 σε 2 μέρη. Αρχικό κείμενο. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό παράγραφος να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος του παραγράφου 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παράγραφος 19 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παράγραφος 23 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παραγραφός 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παραγραφός 27 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Παραγραφός 28 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παραγραφός 32 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παραγραφός 37 αρχικό σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 50 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 53 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 55 υπέρ, να επαληθεύσουμε την 53 μέρος δεύτερο. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτό. Παραγραφός 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Παραγραφός 58 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 66 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 73 υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 77 υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 92 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό παράγραφος 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 94 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας και γίνεται δεκτό. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για ένα ψήφισμα της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων για τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2014. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία expert. Κατά. Θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 1 με ονομαστική ψηφοφορία. Όχι, συγγνώμη. Α, μετά την παράγραφο 1 Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Παράγραφος, ε, τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά δεκτή τροπολογία 4 να επαληθεύσουμε την τροπολογία 2 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας Δεκτή. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Ακόμη λιγότερη. Δεκτή. Παράγραφος 3 αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Το ψήφισμα στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Die haben alle abgestimmt. Ψήφισαν όλοι πέρας γίνεται δέκτη συγχαίρω όλους τους συγητές σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτα έκθεση Κόβατσικ. Η κυρία Πιετικάινεν είναι. Η κυρία Πιέτη